Αν Πρέντα αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Ο κύριος Πρέντα θα μιλήσει πρώτος για τέσσερα λεπτά. Και καλωσορίζω την κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα καταφέραμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συμπεριλαμβανομένης της γενεκτονίας, δηλαδή της φεκαλαιότητας. Θα πρέπει να καταστήσει όλους σαφές ότι ε, τα θέματα αυτά δεν μπορούν να παραμένουν ε, κρυμμένα. Η τελευταία δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ ε, έχει πια ηλικία 6 ετών. Το Συμβούλιο ε, βλέπουμε να αρχίζει να ασχολείται με τα θέματα αυτά τους τελευταίους μήνες και ε, αυτά τα θέματα επίση είναι αντικείμενο διεθνών δικαστηρίων και διεθνών δικών. Να θυμίσω την, το τελευταίο ψήφισμα τη Αφρικανική Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση αυτή επιμένει στην απαράδεκτη κατάσταση και το καθεστώ που είναι απαράδεκτο για τον πληθυσμό του Ρωμά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν οι απαραίτητε προποθέσει για την άριστη λειτουργία του σχετικού δικαστηρίου για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση να αξιολογήσει τι προσπάθειε που καταβαλλόνται εδώ και χρόνια για την προσπάθεια των τρίτων χωρών να ε, συμπληθούν στην ανάλογη σύμβαση και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα δράσης το 2011 για να δούμε πού έχουμε φτάσει ε, ω προ την εφαρμογή ω τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να χαιρετήσω την προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το δικαστήριο σε στι προσπάθειε μετάβαση του 2015. Εδώ πρέπει να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο εξή. Είναι σημαντική και η πρόληψη μετά την, πριν την εκδίκαση μάλλον των σοβαρών εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας είναι σημαντικό να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταβάλει προσπάθειες για να σκεφτεί και να προλάβει όλες αυτές τις καταστάσεις που μπορούν να εγκληθούν σε εγκληματικές συμπεριφορές. Ε, μεγαλύτερη έμφαση στη δράση. Το να αντιδρούμε είναι σημαντικό αλλά πρέπει να γίνεται και σε συνεργασία με τους διεθνούς εταίρους. Εκτιμώ λοιπόν ότι πρέπει να ε, τοποθετηθούμε έντονα στι διμερεί σχέσει μα με τι ενδιαφερόμενε χώρε. Είναι σημαντικό οι διπλωματικέ μα υπηρεσίε να καταλάβουν τι απαραίτητε προσπάθειε εναντί τέτοιου είδου εγκλημάτων. Ο τρίτο άξονα τη έκθεσή μου αφορά την ατιμορρησία των δραστών. Βεβαίω, επικεντρώνουμε στην περίπτωση του Νταέσ, του Άιζη, γιατί η γενοκτονία στο Ιράκ και τη Συρία με την ε, εξάλληψη των μειονοτήτων στην περιοχή είναι έγκλημα αυτή τη οργάνωση. Εδώ λοιπόν δύο επιλογέ έχουμε μπροστά μα. Πρώτα απ' όλα δίωξη ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου ή η θέσπιση ειδικού Διεθνού Δικαστηρίου για το Ιράκ και τη Συρία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη μελέτη αυτών των δύο διαφορετικών επιλογών, διότι το μόνο μόνο που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε είναι η διφορία. Απορρίπτω τα επιχειρήματα που λένε ότι η γεωστρατηγική κατάσταση δεν θα επιτρέψουν ποτέ να περάσουμε το Διεθνέ Δικαστήριο ή να ε, ιδρυθεί ειδικό δικαστήριο. Το γεγονό ότι το Διεθνέ Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία στο Ιράκ και τη Συρία η Ρωσία είναι μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΙΕ, δεν πρέπει να μα σταματήσουν τα στοιχεία αυτά. Χρειάζεται πολιτική τόλμη για να καταδικάσουμε τον Daesh ISIS και να αποκαταστήσουμε τη μνήμη των θυμάτων. Εδώ η ε, διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από τον ΤΑΕΣ συνεχίζονται. Όμω δεν πρέπει να επιτρέψουμε την δημιουργία τέτοιων ανθρωπιστικών κρίσεων από το ΆΕΖΙΣ. Πρέπει να ανακόψουμε την πορεία του ω Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί τον ΟΗΕ και γνωρίζοντα ότι οι δύο τουλάχιστον κάτι η Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο, έχουν αναλάβει ενεργό δράση σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει ο πρωταρχικό στόχο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμμετοχική να οδηγήσει στην καταδίκη των δίμιων αυτών και να φροντίσουμε η ανεξαρτησία της κοινωνίας του Ιράκ και τη Συρία να ενισχυθούν. Θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας για χώρες που έχουν πληγεί μαζικά από την τρομοκρατία του ISIS, αλλά για όλους τους Ευρωπαίους που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία και θέλουν πλέον να υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση. θα πρέπει και τους ξένους μαχητές ISIS και Daesh που θέλουν ανενόχλητοι να επιστρέφουν στη χώρα τους να μην τους αφήσουμε να δρουν ανενόχλητοι. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει ε, πυγμή και αντιμετώπιση, εκδίκαση των περιπτώσεων αυτών στο Διεθνέ Δικαστήριο. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίσει τι πολιτικέ τη ε, στο θέμα αυτό και ευχαριστώ τι πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία του. Λυπούμε που δεν μπορούσαμε να έχουμε ανταλλαγή απόψε. Πολύ σύντομη παρουσίαση. Μόνο αυτό μπορέσαμε να αποσπάσουμε για το θέμα αυτό, αλλά χαίρομαι που βλέπω εδώ την είπατε εκπρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Σας ε, καλωσορίζω όλους. Ε, θα προεδρεύσω μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ όσους ε, έχουν ακόμα την δύναμη να παραμείνουν εδώ στην αίθουσα. Όπως γνωρίζετε, ε, θα ε, ακολουθήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Είχαμε προβλέψει πέντε λεπτά, αλλά ζήτησαν πολύ το λόγο, οπότε έχω δεχτεί 11 ομιλητέ. Θέλω να δώσω την ευκαιρία σε όλου να μιλήσουν. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι και ο εισηγητή ζήτησε όλοι να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Οπότε σας ζητώ Παρακαλώ πολύ περιοριστείτε στο χρόνο το οποίο σας έχω ε, δώσει. Ο κ. Πόσπης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πάρω το λόγο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον, να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα για την έκθεσή του. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε τα εγκλήματα πολέμου, σαφέστατα, και είναι σημαντικό να έχουμε τα κατάλληλα μέσα στα χέρια μας. Θα πρέπει οι, τα όργανα που διαθέτουμε να μπορούν να μας προειδοποιούν έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους εγκλήματα. Θα ήθελα να στηρίξω την ύπαρξη αυτού του ενός τέτοιου μητρώου ας πούμε. Ε, θα θέλαμε επίσης όλο και περισσότερες χώρες να ε, ενταχθούν στο καθεστώς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα πρέπει να οθήσουμε ε, τους εταίρους μας να πάρουν στα σοβαρά αυτό το όργανο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε κυρια Κύριε Βόρντ έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου που εργάστηκαν σε αυτήν την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται ε, και οι συγκρούσει αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Ε, μεταξύ των άλλων θεμάτων τα οποία καλύπτονται από την έκθεση θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών σε ζώνε ε, ε, σύγκρουσης. Οι γυναίκε θα πρέπει να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόληψη ε, των συγκρούσεων και στην στο χτίσιμο της ενίσχυσης και της συμφιλίωσης. Έχω συνεργαστεί με γυναίκες που έχουν ε, στα Δυτικά Βαλκάνια επιζήσει πολέμων ε, και ε, σεξουαλικών επιθέσεων, ιδιαίτερα στο Κωσυφοπαίδιο. Χρόνια μετά οι γυναίκες αυτές ακόμα περιμένουν την απόδοση της δικαιοσύνης και οι ηγέτες μας θα πρέπει να δώσουν αυτή την υποστήριξη πάρα πολλές γυναίκες έχουν επιβιώσει εγκλημάτων πολέμου ε, και ε, δεν έχουν δικαιωθεί. Θα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή τους για να επικρατήσει πραγματική ειρήνη και δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ να τηρείτε το ένα λεπτό. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Να υπάρχει σκληρή τιμωρία και φυσικά να διώκονται οι υπέτειοι. Φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μια πολιτική που να προλαμβάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα. Όσοι είναι υπέτειοι βλέπουν πλέον το τι συμβαίνει στο παρελθόν και αποθρασύνονται. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στην περίπτωση της άρνησης της Γερμανίας να καταβάλει τις γερμανικές αποζημιώσεις προς την Ελλάδα. Παρότι υπάρχει απόφαση από το 1946 ε, της, Συμφωνίας Ειρήνης των Παρισίων, η γερμανική πλευρά αρνείται να καταβάλει τις πολεμικές επανορθώσεις, αρνείται να επιστρέψει το κατοχικό δάνειο, αρνείται να αποζημιώσει τους συγγενείς των θυμάτων για τα εγκλήματα πολέμου που έκαναν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην Ελλάδα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει και πρέπει η γερμανία πραγματικά να καταβάλει τις οφειλές της προς την ελλάδα. να λοιπόν τα μηνύματα που πρέπει να υπάρξουν στα θέματα αυτά. ευχαριστώ. Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια για να καταγγείλουμε και να πάψει ατιμορρησία για κάθε είδου έγκλημα, έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα, έγκλημα πολέμου, γενοκτονία. Δεν μπορούμε ωστόσο να συμμεριστούμε τον κινησμό και την υποκρισία που εμπνέει το ψήφισμα αυτό όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο παραπλανητικό και γεμάτο προκαταλήψει όταν κατανομάζονται χώρες ανάλογα με τα γεωτρατηγικά μας συμφέροντα και τα οικονομικά μας συμφέροντα. Εδώ η οπτική γωνία που ακολουθούμε είναι συγκεκριμένη και χωρίς ε, καμία έκπληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοδική Αραβία, το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά μέλη της δεν κατανομάζονται. Αυτοί που θα έπρεπε να δίνουν ε, ε, το παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο έχουν διαπράξει επικαλότητες κατά των λαών του. Εδώ λοιπόν αυτή η ρητορική υπέρ του Διεθνούς Δικαστηρίου έχει σκοπό να ε, καταβάλει τα κυριαρχά δικαιώματα των ε, λαών και το είδαμε και με την πρόσφατη ιστορία με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γεωκοσλαβία, τα εκατομμύρια ε, θυμάτων και τις τόσες αθώες ζωές που χάθηκαν. Ευχαριστώ πολύ που τήρησατε το χρονικό όριο. Δεν, έχουμε δεν, δεν γίνονται δεκτέ οι μπλε κάρτε, πρόκειται για διαδικασία Η Μπάρμπαρα έχει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτρέπει περισσότερο αυτά τα εγκλήματα και να φροντίζει να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι και με τη βοήθεια του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου. Οι έρευνες πρέπει να συνεχίζονται σε εικαζόμενα εγκλήματα. Θα πρέπει να ξέρουμε πού συντελούνται τα εγκλήματα. Πρόσφατα ε, το κάναμε αυτό για την Ιεμένη. Πρέπει να καταδεικνύονται υπεύθυνοι. Δυστυχώς δεν συμφωνήσαμε ε, σε ε, σχέση με την καταδίκη υπεύθυνων στην Σαουδική Αραβία. Ε, ε, εμείς θέλουμε να ζητήσουμε και ε, ένα ετήσιο κατάλογο περιπτώσεων παραβίασης από τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. κύριο Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε παρά το γεγονό ότι βρισκόμαστε στον 21ο ε, αιώνα και θα περίμενε κανεί τα ήθη του πολέμου να έχουν εξευγενιστεί δυστυχώ ακόμη και σήμερα υπάρχουν εγκλήματα πολέμου εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα και γενοκτονίε. προκειμένου να κάψουν το ηθικό του εχθρού κάποιοι εμπόλεμοι μετέρχονται βασανιστήρια και διάφορε μεθόδου εξευτελισμού και εκφοβισμού του αντιπάλου όπω ε, βιασμού ανδρών και γυναικών σεξουαλική βία κατά των γυναικών ε, ομαδικέ δολοφονίες θρησκευτικών και εθνικών ομάδων και βομβαρδισμούς αμάχων με χημικά όπλα. το άσχημο είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση παρεμβαίνουν και μη κρατικοί φορείς όπως η Boko χαράμ στην Ιγυρία και ο Άισι στο ιράκ και τη συρία που δεν ελέγχονται. για να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση αλλά και η διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει μια στρατηγική η οποία θα προβλέπει την πιθανή εκδήλωση τέτοιων ε, δραστηριοτήτων να τις προλαμβάνει και κυρίω να τιμωρεί άμεσα και πολύ σκληρά αυτού που είναι υπεύθυνοι. όμω για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι αμερόληπτοι και να εφαρμόζονται οι ε, τιμωρίε αυτέ σε όλου όχι όπω η συρία που καταδικάζουμε τι ακρότητε του καθεστώτος Σάσα, αλλά όχι και των αντιπάλων του. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σόιντροβα. να ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πρέντα για την έκθεση. Θα κάνω κάποια σχόλια. Το Σαββατοκυριακό η Συριακή κυβέρνηση απόρριψε την πρόταση για ε, καταδίκη της χρήσης ε, σαρίν ε, που οδήγησε στο θάνατο 8 ανθρώπων η... θεώρησε ότι η, έκθεση, η σχετική έκθεση δεν είναι αξιόπιστη και η Ρωσία είπε ότι αυτό είναι προϊόν χειραγώγησης. Αυτό το καταδικάζω. Η ουδέτερη αυτή έκθεση δεν μπορεί να καταδικάζεται και να απορρίπτεται από την Ρωσία. Γιατί η χρήση του Σαρίν ε, ε υπήρξε και πρέπει τώρα να διερευνηθεί από το δικαστήριο. Επίσης, πολλές φορές σε μειονότητες, σε αγροτικές περιοχές ε, είναι θύματα ε, εγκλημάτων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσάμπας Όγκορ. Ευχαριστώ. Τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συνεχίζουν να διαπράττονται παγκοσμίω Φαίνεται η μακροχρόνια ειρήνη και σταθεροποίηση να είναι κάτι που έχει πετύχει ως όνειρο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή τη στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ε, προλάβει τα δεινά αυτά στον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως ε, βλέπουμε ήδη συνέπειες ε, του τι συμβαίνει γύρω μας στην δική μας κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη μελλοντική πρόληψη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Βλέπουμε ότι χωρίς τη χρήση πολιτικής, στρατιωτικής βίας, στρατιωτικής πυγμής δεν είναι εύκολο να ε, προλάβει κανείς τα εγκλήματα πολέμου μπορεί μόνο μετά από στρατιωτική παρέμβαση επιτόπου να ε, ε, ασκήσει την επουλωτική δράση. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προλάβει εγκλήματα πολέμου, πρέπει να προσφέρει και τα κατάλληλα μέσα, Η ιδάλλως μόνο το ΝΑΤΟ θα αναλάβει αυτό το βάρος και την ευθύνη. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Στάνισλαφ Μπόλτσακ και μετά η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι πεπισμένο ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένη τη γενοκτονία, πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτηση και πολύ κακό συζητούνται τόσο αργά σήμερα. Εκτιμώ το γεγονό ότι η έκθεση του κυρίου Πρέντα είναι πλήρη και η πρόληψη, όπω ε, αναφέρθηκε, αλλά και η αντιμετώπιση τη είναι θεμελιώδου σημασία. Εδώ υπάρχει και μια νομική πτυχή όμω την οποία θέλω να επισημάνω. θέμα διεθνούς δικαίου που αφορά και την περίπτωση της λύθης για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα απόκρυψης τέτοιων εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κοντά της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να υπάρχει και διάρκεια στο κατά πόσο, στο, ε, να υπάρχει μια συγκεκριμένη διάρκεια για την περίοδο δίωξη των ε, υπευθύνων και των αυτούργων, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον κάποια στιγμή στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση στα πλαίσια τη σύντομη παρουσίαση και τώρα ο λόγος στην ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο, τον κύριο Πρέντα, για τη δουλειά του, για την έκθεση αυτή. Να πω, Πρόεδρε, ότι έχω συνηθίσει τις νυχτερινές ολομέλειες ε, του Στρασβουργού αν και ε, δεν μου φαίνεται πολύ λογικό να καθυστερούμε τουλάχιστον δύο ώρες αύριο. Επίσης θα είμαι εδώ το βράδυ, στην ώρα μου, αλλά καλό θα ήταν να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση του χρόνου. Η δουλειά μας για να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπότητα και εγκλήματο κατά της ανθρωπότητας. Είναι και θέμα του κατά πόσον προστατεύουμε τη δική, τα δικά μας συμφέροντα με το επόμενο έγκλημα πολέμου, την επόμενη σύγκρουση να οδηγεί σε νέο πόλεμο με περισσότερε παραβιάσει. Οι συγκρούσει και οι εχθροπραξίε κάνουν τη συμφιλίωση και την ειρήνευση πολύ ε, δύσκολη και δύσκολη τη δουλειά μας, ιδίω για τη φάση της ε, αποκατάστασης μετά. Η καχυποψία, η καταστροφή της κοινωνίας, ε, οι πληγές μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να επουλωθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους η ευθύνη μα να προστατεύσουμε και να προλάβουμε τις φρικαλαιότητε, όλα αυτά είναι μέρος όλων των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Συμφωνώ κατά πολύ με την έκθεσή σα, που δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και σε αυτέ τι εβδομάδε ακριβώ. Θεσπίσαμε ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που καταγράφει και τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Οι ομάδε μα και οι διπλωματικέ μα αποστολέ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν εδώ για την πρόληψη αλλά και με τι αντιληπτικέ αρχέ τη ε, ενδιαφερόμενε χώρε και την κατάλληλη εκπαίδευσή του πρέπει να συνεργαστούμε. Με τα χαράς βλέπω ότι η εκθεσή σας καταγράφει και άλλα σημαντικά στοιχεία του, της δουλειάς που κάνουμε τώρα, όπως τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική βία. Μόλις πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολήθηκε με την απόκριση σε τέτοιου είδου μορφέ βία, με 3,5 εκατομμύρια γυναίκε, άντρε και παιδιά να είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Το τελευταίο πακέτο για τη στήριξη των ε, σύρων προσφύγων ε, προέβλεπε την προστασία από τέτοιε μορφέ σεξουαλική βία για 700.000 Σύρου εντό και εκτό χώρα. Όμω για την πρόληψη ξέρουμε ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα συμβαίνουν σήμερα και εμεί έχουμε καθήκον να ασχοληθούμε και με τι συνέπειε. Η δικαιοσύνη είναι το μόνο δραστικό μέτρο και η μόνη βιώσιμη απόκριση σε τέτοιου είδου μορφέ βία. Η ατιμορρησία δημιουργεί περισσότερο μίσο, προξενεί περισσότερο πόνο και τη διάθεση εκδίκηση. Η απόδοση δικαιοσύνη είναι ο μόνο τρόπο για να υπάρξει συμφιλίωση και μακροπρόθεσμη ε, βιώσιμη ειρήνη. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να συνδυάσουμε διαφορετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα την ποινική δικαιοσύνη, τις αποζημιώσεις, την ε, θεσμική μεταρρύθμιση. Να αναφέρω μερικέ περιπτώσει όπου εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να προλάβουμε την ατιμορρυσία, να την αντιμετωπίσουμε και να αποδώσουμε δικαιοσύνη στη Συρία. Ε, θέλουμε να υπάρξει διεθνή και αμερόληπτο μηχανισμό απόδοση δικαιοσύνη που να λειτουργήσει το δυνατόν πιο άμεσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί κονδύλια για να στηρίξει το μηχανισμό αυτό με 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι τα κάτι μέλη έχουν αναλάβει το δικό του μερίδιο και υπολογίζω σε αυτά ε, και στη στήριξή του για να έχουμε ίσω και μεγαλύτερη στήριξη από την πλευρά των εθνικών κρατών στο Ιράκ, καθώ απελευθερώνονται και άλλε περιοχέ από τον Ντάεσ Άιζη, πρέπει να αποτιμήσουμε τα κλίματα πολέμου και τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν δεσμεύσει από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ και την τοπική κυβέρνηση του Κουρδιστάν να γίνουν ασφαλεί ανακριτικέ έρευνε ε, για το τι εγκλήματα έχουν διαπράξει οι Ιρακινέ δυνάμει. Ε, στη Συρία και στο Ιράκ πέρσι είχαμε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΙΕ για να δημιουργηθεί επιτροπή, επιτροπή και για την περίπτωση του Μπουρούντι και στηρίζουμε και την ανάλογη απόφαση της Γενέβη του περασμένου μήνα να υπάρξει ένας μηχανισμός ε, για την διερεύνηση παρομοίων εγκλημάτων στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την αναγνώριση της πολύ εντατικής μας δουλειάς και την στήριξη του διεθνού Δικαστηρίου ε, για τα εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Από το 2000 έχουμε 30 εκατομμύρια ευρώ ως άμεση στήριξη του δικαστηρίου αυτού και το, περασμένο, το περασμένο Σάββατο προβλήθηκαν 15 χρόνια. Μάλλον αποτιμήσαμε τα 15 χρόνια λειτουργίας του δικαστηρίου με την, ε, με την οικουμενική ε, δήλωση για τους Ρωμά να εγκρίνεται. Επίσης πολλά αφρικανικά κράτη, η Γκάμπια, η Νότια Αφρική και το Μπουρούντι έχουν δεχτεί το καθεστώς δικαστηρίου δυστυχώς ε, και ευτυχώς ανακάλυψαν προηγούμενες αποφάσεις εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η σχετική δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί. Κοιτάζουμε πώς να Η σύμβαση της Ρώμης επίσης πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και να ε, ε, εγκριθεί ε, παγκοσμίως από όλα τα κράτη. Εδώ οι προσπάθειες λοιπόν συνεχίζονται. Πρέπει να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δεν, υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία για την ε, στήριξη της πολυμερούς διακυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κάτω δικαίου με ισχυρούς φορείς και θεσμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να είναι αξιόπιτος, αξιόπιστος, αναγκαίος και σταθερός σύμμαχος του ΟΗΕ και για όλους όσοι πιστεύουν ότι στη βία πρέπει να απαντούμε με δικαιοσύνη και συμφιλίωση. Τη δουλειά αυτή θέλουμε να τη συνεχίσουμε μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο, στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μογκερίνη. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση των δύο ωρών. Το πρώτο μισάωρο αφιερώθηκε στη μνήμη της Σιμών Βέιλ και μετά βέβαια είχαμε κι εμείς μια ευθύνη στις καθυστερήσεις. Ε, σας υπόσχομαι την επόμενη φορά να αφιερώνουμε μόνο πέντε λεπτά στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και ευχαριστώ πολύ που μας το υποδείξατε.